Eh, Καλημέρα σε όλους, αγαπητοί συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε τις εργασίες μας από το σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε στις 10 ε, Ιουλίου. Και έχει... Τους ενιαίους κανόνες ε, και την ε, ενιαία διαδικασία για χρηματοπιστωτικά αισθητήτα και οργανισμούς και επενδυτικούς οργανισμούς για ένα ενιαίο ταμείο εξυγίασης και ενιαίο μηχανισμό εποπτείας. Θα δώσω το λόγο καταρχήν στην εισηγητριά μας, την κυρία Φερέιρα, εκ μέρους των σοσιαλιστών. Έλίζα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το, το κείμενο, το έγγραφο που έχουμε στην ημερήσια διάταξή μας είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο από πολλές απόψεις και σε πολλά επίπεδα. Και κάνει ουσιαστικά ένα βήμα επιπλέον σε όλο αυτό το αρχιτεκτόνημα της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουν το κείμενο αυτό. Εγώ θα παριθμίσω τα βασικά μου στοιχεία. Είχαμε μία πρώτη άτυπη συνάντηση. Όλοι οι εισηγητές που συμμετέχουν στη συζήτηση και στη διαμόρφωση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Ενίο μηχανισμό εξυγίανσης. Και μπορώ να σας μεταφέρω τις βασικές απόψεις από τις συζητήσεις. Κανένας δεν θεωρεί ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη νομική βάση πάνω στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριξε την, της, την πρότασή της. Όλοι θεωρούμε λοιπόν ότι η νομική βάση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σωστή. Επίσης, όλοι οι ευρωβουλευτές που συμμετείχαν στην ομάδα αυτή εξέφρασαν την θέλησή τους να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό στη διαμόρφωση τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για, τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίασης. Γιατί αυτό ο μηχανισμό είναι ε, ζωτική σημασίας. Γιατί ήδη την περασμένη εβδομάδα εγκρίναμε τον ενιαίο υποπτικό μηχανισμό. Και από τη στιγμή που έχουμε μια ενιαία υποπτία για τις χώρες της Ευρωζώνης και για τις χώρες που εθελοντικά θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το μηχανισμό, δεν έχει νόημα να έχουμε από τη μία μία ενιαία υποπτία και από την άλλη οι χρηματοπιστωτικές ε, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να υπάγονται μόνο στα, στις εθνικές αρχές γιατί όλη η αρχιτεκτονική του συστήματος ε, προϋποθέτει μία διαλειτουργικότητα των διαφόρων ε, σημείων και των διαφόρων πυλώνων και ένα συντονισμό μεταξύ τους. Με αυτή τη λογική θέλουμε να επισπεύσουμε τη διαδικασία και περιμένουμε από το Συμβούλιο να δείξει το ίδιο μέλημα και την ίδια σπουδή. Θεωρούμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, παρά τις ε, βελτιώσεις που επιδέχεται και τις ε, τροπολογίες, ως προς την βασική της ρεχοκοκαλιά και το βασικό της σκελετό χρήζει επιδοκιμασίας και έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα έχουμε κάποιες λεπτομέρειες. Μία από αυτές αφορούν το γεγονός ότι δεν ε, εργαζόμαστε παράλληλα με την οδηγία RRD, δηλαδή την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίαση των τραπεζών που δημιουργεί ένα ενιαίο ομοιόμορφο νομικό πλαίσιο για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ενώ προχωρούμε με τον ενιαίο μηχανισμό ε, εξυγίασης ε, για τις χώρες της Ευρωζώνης ε, και τις χώρες που και ο Θεός ενταχθούν, δεν έχουμε ταυτόχρονα και πολλές παράλληλες, πάλι παράλληλη πρόοδο στην οδηγία για την ανάκαψη και εξυγίαση τραπεζών. Ένα τμήμα του κειμένου του ενιαίου μηχανισμού εξυγίασης μένει εκρεμές εν αναμονή Τη έκβαση των διαπραγματεύσεων που συνεχίζονται ακόμη μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξηγήση των τραπεζών, την RRD. Θέλω αυτό να ρωτήσω τους συναδέλφους αν έχουν την αίσθηση και αν συμφωνούν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε μια νέα πλατφόρμα με μια νέα νομική βάση και αν θεωρείτε ότι θα πρέπει να έχουμε στην σχέση μεταξύ των κανόνων της ε, εξηγήσης των τραπεζών για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και των κανόνων που ισχύουν ιδιαίτερα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εμπίπτουν στην Τραπεζική Ένωση. Επίσης θα πρέπει η Γραμματεία να μας υπεβεβαιώσει ποια άρθρα παραμένουν εκκρεμοί ενώσο αναμένουν, αναμένουμε τις διαπραγματεύσεις ε, της για την ε, εξηγήση και την ανάκαμψη των τραπεζών. μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που κατά τη γνώμη μας χαρίζουν περαιτέρω διευκρίνησης. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ε, αρμοδιότητες αυτού του συμβουλίου, του board ή του οργάνου που σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιληφθεί της εξυγίασης στα πλαίσια της Τραπεζικής Ένωσης. Και ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί θεωρούμε ότι θεσμικά και νομικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει το λόγο στις αποφάσεις. Αλλά σε ό,τι αφορά τις, ε, το νομικό κείμενο, θα πρέπει να αποφεύγουμε παρερμηνίε και να έχουμε σωστή στο συντονισμό και συνοχή μεταξύ του νέου αυτού του Board και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό είναι ένα θέμα που συνδέεται άρρηκτα με το θέμα της ε, δημόσιας παρουσίας των λογαριασμών και το θέμα της, το θέμα της Είναι μια λειτουργία πολύ σημαντική και πιστεύουμε ότι στο νομικό κείμενο θα πρέπει να γίνει ένας παραλληλισμός μεταξύ του αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων του Κοινοβουλίου και των λιπόθεσμικών οργάνων σε ό,τι αφορά τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη, στο διορισμό του εκτελεστικού υπευθύνου της αρχής της εξυγίασης και θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας παραλληλισμός σε ό,τι αφορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των στοιχείων ε, της ε, δημόσιας παρουσίασης των λογαριασμών με αυτό που πετύχαμε στην εποπτεία και αυτό που θα δημιουργήσουμε τώρα στη διαδικασία εξυγίανσης. Ιδιαίτερα δηλαδή στο διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή. Είπαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θέλουμε μια ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων και είναι σημαντικό και το θέμα της παρουσίας, της συμμετοχής του. Γιατί το έργο του είναι πολύ σημαντικό. Θα είναι ο διευθυντής μιας πολύ σημαντικής ε, αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ αναφέρω τις αδρές γραμμές κάποιων ε, σημαντικών σημείων. Δεν πρόκειται να απορριθμίσω όλες τις λεπτομέρειες του κειμένου. Ε, δύο άλλα θέματα που είναι σημαντικά ε, και θα τα αναφέρω τώρα γιατί περιμένω με ανυπομονησία τις απόψεις του συναδέρφου, των συναδέρφων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, προτιμάει τους καταθέτες στην ιεράρχηση του Μπέιλιν της, της διάσωσης με ίδια μέσα δηλαδή. Θέλουμε να προτιμησιακή μεταχείριση ε, σε ό,τι αφορά τις επιλέξιμες καταθέσεις. Αυτό το θέμα είναι φλέγον, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών και θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα του bail-in ε, και το κατά πόσο θα πλήξει αυτό τις εγγυήσεις καταθέσεων. Αυτό είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα γιατί η χρήση της εγγύης καταθέσεων σε, στις διάφορες προσπάθειες ανάκαμψης μιας τράπεζας μπορεί να καταστούν μη βιώσιμες. Ιδιαίτερα αν δεν ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια. Σε αυτό το θέμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατράνωσε με σαφήνεια τη θέση του. Και θα, ίσως θα χρειαστεί να τα διαμορφώσουμε κάπως περαιτέρω στις ε, διαπραγματεύσεις. Τέλος, από τη στιγμή που θα έχουμε ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ανέκαθεν ε, υπέρ ε, της ε, οδηγίας για την εξυγίαση των τραπεζών, θεωρούμε ότι τα κονδύλια που θα χρησιμοποιηθούν για παρέμβαση σε περίπτωση πτώχευσης ή διαδικασίας ε, εκαθάρισης μάλλον ή εξυγίανσης μιας τράπεζας τα κονδύλια αυτά θα πρέπει να είναι ιδιωτικά, να χρηματοδοτούνται από την ίδια την τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ανέκαθεν υπέρ αυτής της άποψης. Οπότε η πρόταση για ένα κοινό ταμείο και ένα ταμείο που θα χρηματοδοτείται από τις τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ανάλογα με τους κινδύνους που εισαγάγουν στο σύστημα, πιστεύουμε ότι αυτή η αρχή είναι η σωστή. Αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε πως ειδικά στην πρώτη περίοδο της λειτουργίας αυτού του συστήματος και όσο διαμορφώνεται αυτό το ταμείο θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο είναι χρήσιμο να έχουμε ήδη κάποια κονδύλια και πιστώσεις ε, που θα εγγυώνται την σταθερότητα αυτού του ταμείου από την ε, αρχή της λειτουργίας του, όπως είχαμε προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο κείμενό μας το 2010. ιδιαίτερα ο συνδυασμός του Ταμείου με το μηχανισμό σταθερότητας και το, μηχανισμό με το σύστημα χρηματοπιστωτικής ε, σταθερότητας. Είναι σημαντικό αυτό για να έχουμε ένα συντονισμό της παρέμβασης και όχι ακανόνιστες παρεμβάσεις ή άτακτες παρεμβάσεις σε τράπεζες που βρίσκονται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης ε, τακτικής εξηγίασης, συντεταγμένης εξηγίασης. Αυτά λοιπόν ήταν τα δύο πιο στεναρά θέματα σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία της παρέμβασης. Αλλά σε γενικές γραμμές το κείμενο είναι καλό και είναι ένα κείμενο που χρειαζόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση βασικός πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης για να υλοποιήσουμε τους τρεις πρωταρχικού μας στόχους. Την καλύτερη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την προστασία των φορολογουμένων που μέχρι στιγμής ήταν τα θύματα των προβλημάτων των τραπεζών και η προστασία των καταναλωτών. Αυτοί είναι οι τρεις πρωταρχικοί μα στόχοι, η προστασία των καταθετών δηλαδή. Και είμαστε πεπισμένοι ότι με αυτά τα τρία στοιχεία, με την υλοποίηση αυτών των στόχων, η τράπεζα θα ανακτήσει την πρωταρχική της λειτουργία, που είναι να μετατρέψει τις καταθέσεις σε επιστώσεις στην πραγματική οικονομία. Γιατί έτσι θα τονώσει την πραγματική οικονομία και θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διέλθει από αυτή την παρατεταμένη κρίση την οποία βιώνει. Περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις θέλω να συνεργαστούμε με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρώ ότι υπάρχει συνεργάσιμο πνεύμα μεταξύ των πολιτικών ομάδων και ισχυρή βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιταχύνει στο έπακρο τις διαδικασίες ε, διατρανώντας τη θέση του για αυτό το νομοθετικό κείμενο. Και ευελπιστώ ότι και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα συμμερίζονται αυτό το πνεύμα για την ταχεία πρόθεση των εργασιών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Ελίσσα. Εκ μέρους του ΕΛΚ τώρα και λήψη της σκιώδους συγγήτριας, της κυρίας Βόρτμαν Κόλ, θα δώσω το λόγο στον συντονιστή μας, τον κύριο Κοζές. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως το είπατε κι εσείς, θα μιλήσω εξ ονόματος κυρίας Βόρτμαν Κόλ, η οποία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έρθει εξαιτία μιας διαδήλωσης μεγάλης που γίνεται στη χώρα Τη Σα ζητά συγγνώμη για την απουσία. Επομένως θα εκφράσω τις δικές της αποφά, τις δικές της προτάσεις εφόσον είναι σκιώδης ε, εισηγήτρια για το ζήτημα αυτό. Μας λέει λοιπόν η συναδελφός μας ότι καταφέραμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα την προηγούμενη εβδομάδα δημιουργώντας το νέο αυτό συμβούλιο και τη νέα δυνατότητα εποπτείας πλέον που θα έχει το, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να καταφέρουμε να κτίσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στο τραπεζικό σύστημα. Θα πρέπει να καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες, να ακολουθήσουμε ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα προκειμένου να τηρήσουμε την προθεσμία της θέσης ισχύω της 1ης Ιανουαρίου του 2010. 2015. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βασιστούμε στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό για τον οποίο εισηγείται την η κυρία Τάισεν προκειμένου να καταφέρουμε να διαχειριστούμε καλύτερα τις κρίσεις στο μέλλον κυρίως μέσω του ε, νέου συστήματος ε, ενιαίας εξυγίανσης των τραπεζών θα πρέπει να δώσουμε στη δυνατότητα, την, στην αρχή εξυγένσης ε, στις δυνατότητες να αναλάβει δράση πολύ γρήγορα, να μπορεί να προλαβαίνει τις ε, κρίσεις κάθε φορά που μια τράπεζα παρουσιάζει προβληματικά στοιχεία ή διανύει μια κρίση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τα χρήματα των φορολογωμένων και των καταθετών και να καταφέρουμε να προλάβουμε τις ζημίες που προκαλούνται στην πραγματική οικονομία. Γι' αυτό το λόγο, κυρία Βόρτμαν Κόλ υποστηρίζει την φιλόδοξη γραμμή της πρότασης του κυρίου Μισελ Μπαρνιέ, μολονότι ε, επιδέχονται ακόμα κάποιε βελτιώσει ή πρέπει να συζητηθούν κάποιε λεπτομέρειε. Η κυρία Βόρτμαν Κόλ θα ήθελε καταρχά να αναφερθεί στα εξή σημεία. Να αναφερθούμε λίγο περισσότερο στην ε, ε, θέση που θα πρέπει να έχει σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Συμβούλιο Αυτοεξυγίανση. Θα πρέπει να υπάρχει μια εξισορρόπηση αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στις δύο, στα δύο θεσμικά όργανα θα πρέπει το Συμβούλιο, μάλλον θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το Συμβούλιο να καταφέρει να έχει περισσότερες αρμοδιότητες για την εξυγίανση, αλλά ενδεχομένως να πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο αυτό το ενδεχόμενο. Επίσης χρειαζόμαστε ένα ενιαίο ταμείο εξυγίανσης των τραπεζών, προκειμένου να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις κρίσεις. Ενδεχομένως θα χρειαστεί πολλής χρόνος για να δημιουργηθεί το ταμείο αυτό, πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ιδιωτικός να χρηματοδοτήσει το ταμείο αυτό, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναλύσουμε όλες τις δυνατές πιθανότητες που θα έχουμε, δυνατότητες που θα έχουμε, προκειμένου να δημιουργηθεί το ταχύτερο δυνατό το ταμείο αυτό. Η δημοκρατική εποπτεία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις τράπεζες αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αναλύσαμε πολύ το σύστημα της ενιαίας εποπτείας. Νομίζω ότι μπορούμε να επιφέρουμε ακόμα κάποιες βελτιώσεις, όπως για παράδειγμα ο διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή του Συμβουλίου του Board Εξυγίανσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορεί να αναλαμβάνει πιο έντονη δράση όσον αφορά το ενιαίο αυτό ταμείο εξυγίανση τραπεζών και θέλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που μας δίνονται από τη συνθήκη. Θα θέλαμε ωστόσο να πούμε ότι Θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ φιλόδοξοι με, την, ε, με το νέο πλαίσιο εξυγίανση των τραπεζών που δημιουργείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε σε αυτό το πλαίσιο να εντάξουμε και μία ρήτρα αναθεώρηση. Αυτέ είναι οι προτάσει και οι παρατηρήσει που είχε να κάνει η κυρία Βόρτμαν Κόλ. Τώρα εκ μέρου των φιλελευθέρων, η κυρία Γκουλάρη έχει το λόγο. Ε, σε ευχαριστώ, Πάμπλο. Έχουμε την εντύπωση ότι βλέπουμε εδώ πέρα να, να δημιουργείται από την αρχή ένα ολόκληρο σύστημα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι θα καταφέρουμε να εργαστούμε πάρα πολύ καλά, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε την Ολίζα, την Κορίν Βόρτμαντ Κόλ, καθώς επίσης και άλλους συναδέλφους που είχαν εργαστεί και για το Six Pack. Νομίζω ότι όντω πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Πρέπει όντω να δημιουργηθεί το ενίο αυτό Ταμείο Εξυγένση των Τραπεζών. Νομίζω ότι ε, είναι το τελευταίο σκέλο μια μεγάλη εργασία που μα έχει απασχολήσει από την αρχή τη νομοθετική αυτή θητεία. Θα πρέπει να καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο και γι' αυτό το λόγο λέω ότι θα πρέπει ενδεχομένω να έχουμε μια ρήτρα αναθεώρηση, όχι για να ξαναδημιουργήσουμε ένα νέο κείμενο στο μέλλον για να καταφέρουμε τώρα να προχωρήσουμε γρήγορα και να μπορέσουμε να επιφέρουμε κάποιες βελτιώσεις εφόσον χρειαστούν στο μέλλον. Συμφωνώ με πάρα πολλά πράγματα με τα οποία υπόθηκαν όσον αφορά το συντονισμό με το... για το Συμβούλιο αυτό εξυγίανσης. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ καλή εργασία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα έχουμε δύο ουσιαστικά αρχές οι οποίες θα επεμβαίνουν η μία μετά την άλλη οι οποίες έχουν μια διαφορετική σύνθεση, έχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες πολλές φορές, διαφορετικές προσεγγίσεις και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο που μιλάμε για πάρα πολύ σοβαρά πράγματα και ενδεχομένω να μιλάμε για το κλείσιμο μιας τράπεζας και είδαμε στα πρόσφατα παραδείγματα που είδαμε στο Βέλγιο ή στην Γαλλία ή στις κάτω χώρες από την αρχή της κρίσης ότι υπάρχουν όντως κάποια διασυνοριακά ζητήματα τα οποία κάνουν τα πράγματα ακόμα πιο πολύπλοκα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να εργαστούμε ακόμα περισσότερο για αυτό το ζήτημα της εξυγίανσης των τραπεζών. Κάποια πιο τεχνικά ζητήματα, η Επιτροπή αναφέρεται σε μία αρχή επιβολής κανόνων όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. Πρέπει σαφώ να μα απασχολήσει αυτό γιατί αφορά την πολιτική ανταγωνισμού. Πρέπει να δούμε επίση ε, πώ θα καταφέρουμε να λαμβάνουμε πολύ γρήγορα κάποιε αποφάσει όσον αφορά τι κρατικέ αυτέ ενισχύσει που ακολουθούν διαφορετικό, πιο αργό χρονοδιάγραμμα. Και επίση, αν ένα κράτο αποφασίσει να εξέλθει από το σύστημα του ενιαίου υποπτικού μηχανισμού ή από το σύστημα της εξυγίανσης των τραπεζών, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα τα οποία δόθηκαν από το κράτος αυτός, αυτό θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο μέλλον. Δηλαδή να μην εξαφανιστεί η χρηματοδότηση του κράτους αυτού από τη μία μέρα στην άλλη, μόνο και μόνο επειδή θα επέλθει μια κάποια αλλαγή θα αποχωρήσει από το σύστημα. Αυτό το είχα πει και όταν συζητούσαμε και τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις ε, οι οποίες όμως να μπορούν να τηρηθούν και στο μέλλον, να μην ε, ανακαλούνται οι αποφάσεις αυτές πολύ εύκολα από τη μία μέρα στην άλλη. Με την ε, βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε εύκολα μία λύση για να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε το συντομότερο δυνατό τα μέτρα τα οποία έχουμε εγκρίνει. το λόγο Λάμπερτ λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Γκίγκολτ. Δεν είμαι ο κύριος Λάμπερτ, αλλά δεν κάνει μεγάλη διαφορά. Καταρχάς, να μιλήσω γερμανικά. Θα ήθελα από πλευρά μα να παρουσιάσω κάποια κεντρικά σημεία. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια κοινή υπηρεσία εξυγίανση και ένα σχετικό ταμείο για τη δημιουργία ενός σχετικού ταμείου, τονίζοντας το ένα ενιαίο κοινό ταμείο, θεωρώ και θεωρούμε ότι είναι πραγματικά το σωστό, η σωστή κατεύθυνση. Και αυτό γιατί. Γιατί σε κάθε κράτος μέλος υπάρχει μία θα, σε περίπτωση που ιδρύονταν μία ξεχωριστή υπηρεσία, ξεχωριστό ταμείο ανακρατός μέλος, δεν θα ήταν αποτελεσματικό το σύστημα. Είναι παράλογη η πρόταση σε χώρες που είναι μικρές σχετικά να υπάρχει ένα ξεχωριστό ταμείο και ένας ξεχωριστό, μια ξεχωριστή υπηρεσία εξυγένσης. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει απαραίτητη εμπειρία για να προβούν σε εξυγίανση σε περίπτωση που χρειαστεί. Το πρόβλημα θα είναι σε περίπτωση που δημιουργηθούν τελικά εθνικά συστήματα, είναι τελικά ο φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει το λογαριασμό. Για παράδειγμα, στο Μόναχο να υπάρχει, αν υπήρχε σχετικός μηχανισμός, υπηρεσία, ταμείο εξυγίανσης, θα έχει προϋπολογισμό ανάλογο με αυτό κάποιων κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει νόημα λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο. Σκοπό μα θα πρέπει να είναι η Τραπεζική Ένωση. Σε μια Τραπεζική Ένωση θα πρέπει να υπάρχει και το Ταμείο και η Υπηρεσία Εξυγίανση. Δεν έχει νόημα να γίνει διάκριση μεταξύ μεγάλων και μικρών τραπεζών, γιατί και σε μικρέ τράπεζε δεν θα έχει η ανάλογη υπηρεσία Εξυγίανση την εμπειρία προκειμένου να προβεί σε μια εθνική εθνικού επίπεδου εξυγίανση. Και αυτό τι σημαίνει ότι αν δεν υπάρξει μια υπηρεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εξυγίανση των τραπεζών, θα υπονομεύσουμε ε, την ε, τραπεζική εποπτεία. Και δεν είναι λογικό να δίνουμε την εξουσία της εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά να μην αναλαμβάνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ευθύνη. Είναι κατά της αρχής αυτής. Ότι θα πρέπει πάντα να είναι στα ίδια χέρια η εποπτεία, η εξουσία αλλά και η ευθύνη. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχει νόημα στο να υπάρχει ένα δίκτυο εθνικών υπηρεσίων, εθνικών ταμείων. Χρησιμοποιούνται διάφορα νομικίστικα επιχειρήματα. Η δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα για τις περιπτώσεις ε, short selling ε, ανοιχτών πάνε προς την κατεύθυνση αυτή. Και είναι σαφές, σαφές ότι χωρίς ε, αλλαγή και τροποποίηση των συνθήκων είναι δυνατόν να δημιουργηθεί το Ταμείο Εξυγίανσης και στην υπόθεση Μυρώνη, από ό,τι φαίνεται και ο Ζαν Πολ και η Σίλβη τσακώνονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την νομική υπηρεσία. Γιατί έχουν ανακηρύξει εντεκάτη εντολή την υπόθεση Μερώνη. Την ευρωπαϊκή πεποίθηση, την ερμηνεία από πλευράς της νομικής υπηρεσίας ε, της υπόθεσης αυτής. Επιτρέπατε μεταβίβαση τέτοιων ευθυνών σε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία. Πρέπει να υπάρχουν οι σωστοί όροι. Ο Γενικός εισαγγελία δηλώνει ότι βάσει του άρθρου 352 μπορούμε να πάμε πολύ παραπέρα σε ό,τι αφορά την ίδρυση νέων υπηρεσιών και νέων αρμοδιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με δυνατότητα λήψη αποφάσεων. Αυτό δεν θα πρέπει να το αγνοήσουμε. Ξέρουμε ότι βρισκόμαστε. Πόσο δύσκολο θα είναι ένα, να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό συνέδριο και πόσο δύσκολο θα είναι να εφαρμοστούν τα αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την, υπηρεσία, την οδηγία για τις υπηρεσίες. Θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά. Και την έκθεση αυτή. Να αναφέρουμε στην έκθεση κάπου, κάποια στιγμή, ότι είναι ανοησίε αυτά σε ό,τι αφορά την υπόθεση Μυρώνη. Την δεκαετία του 60 είχε κάποια διαφορετική σημασία. Τα πράγματα όμως διαφέρουν πλέον και αυτό το διευκρινίζει ο Γενικός Εισαγγελέας του Λουξεμβούργου. Αν ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αποφασίσουν να μεταφέρουν αρμοδιότητες σε Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, διαφέρουν τα πράγματα. Ελπίζω λοιπόν να ακολουθήσει την κατεύθυνση αυτή το ΔΕΚ προκειμένου να μπορέσουμε να το επιλύσουμε επιτέλους αυτό το πρόβλημα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί? Γιατί το θέμα το οποίο ανακύπτει και το ερώτημα που τίθεται προς την κοινή αρχή ε, επιτήρησης εποπτείας των ε, τραπεζών είναι ποιος είναι ο ανασταλτικός μηχανισμός, ποιο είναι το backstop σε ό,τι αφορά τους ισολογισμούς. Αν δεν υπάρχει αποτελεσματικός ανασταλτικός μηχανισμός, ενδεχομένως η ΑΕΚΤ λόγω φόβου αντίδρασης των αγορών να μην κάνει ένα σοβαρό stress test. Αυτό δεν θα πρέπει να το κάνουμε στον φορολογούμενο τη στιγμή που θέλουμε να κάνουμε τέτοιες, τέτοια μεταφορά ε, αρμοδιοτήτων σε Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή Τραπεζών. Θα πρέπει να μεταφερθεί και η ευθύνη δεν μπορούμε να κάνουμε ένα stress test το οποίο δεν θα είναι σωστό, δεν θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει σχετική πρόταση και αυτό το Ταμείο ε, Ευρωπαϊκής Εξυγίανσης που θα μπορεί να κάνει επαναεπένδυση στην αγορά θα πρέπει να μπορεί να είναι λειτουργικό και θα πρέπει στο πλαίσιο των εργασιών μας να συζητήσουμε προκειμένου αυτό το ταμείο να έχει τη δυνατότητα σε περίπτωση αμφιβολιών να επιλύσει προβλήματα. Καταρχάς λοιπόν θα πρέπει να έχει σωστή χρηματοδότηση, θα πρέπει τελικά να είναι υπεύθυνος ε, ο τραπεζικό τομέα στην τελική ανάλυση και κατά τρίτον να είμαστε τόσο γρήγοροι ώστε εγκαίρω να τεθεί σε εφαρμογή ο μηχανισμό αυτό, γιατί οποιαδήποτε καθυστέρηση θα είναι πραγματικά ανεύθυνη γιατί ουσιαστικά θα υποσκάψουμε την Ευρωπαϊκή Υποπτική Αρχή. Και δύο τελευταίε παρατηρήσει εν συντομία. καταρχά, ε, σε, ό,τι αφορά την ασφάλεια των Ιδρυμάτων στην ε, ε, Γερμανία. Ανησυχεί πολλού αυτό το θέμα δεν θα πρέπει να ισχύει εξαίρεση. Θα πρέπει να έχει δυνατότητα αυτοεξυγίανσης πρακτικά. Και να ευνοείται το σύστημα αυτό όπως ακριβώς ευνοείται το γερμανικό σύστημα εξυγίανσης όπου οι, τα ταμιευτήρια πληρώνουν λιγότερο κόστος, μικρότερα τέλη γιατί έχουν μεγαλύτερες ε, αποδόσεις όπως την έκθεση Πέτερ Ζήμουνς. Να μην υπάρχουν λοιπόν εξαιρέσεις, αλλά να υπάρχει μια διασφάλιση στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό θα εξυπηρετήσει καλύτερα τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες Σωματείων και τις, ε, τα Μιευτήρια. Και ένα τελευταίο θέμα που με ανησυχεί ιδιαίτερος στο Συμβούλιο στην οδηγία για την εξυγίνηση στο άρθρο 72.2, στο συμβαστικό του κείμενο, προβλέπει μία εξαίρεση που θεωρώ ότι κανείς δεν την έχει δώσει τη σωστή σημασία. Τι αναφέρει, ότι πριν ε, αναφερθεί το 8% της συμμετοχής των πιστωτών κτλ, ότι πριν ε, θα, θα, είναι, θα υπάρχει δυνατότητα κρατικών ε, επιδοτήσεων. Σας παρακαλώ κοιτάξτε αυτό το άρθρο 72.2. Ιδιαίτερα εσέ, συνάδελφε Γκούναρ Χουικμαρκ, δεν είναι ε, αποδεκτό οι τράπεζες ε, που έχουν προβλήματα να μπορούν να έχουν επιδοτήσεις κρατικές, χωρίς όρια. Αυτό στα πλαίσια συμβιβασμού προσθέθηκε από πλευρά του Συμβουλίου. Θεωρώ ότι είναι αντιφατικό αυτό με την αρχή ότι και οι τράπεζες θα πρέπει να καλούνται να πληρούν τους λογαριασμούς τους η συμμετοχή των πιστωτών θα πρέπει να γίνεται πριν τις, τις κρατικές επιδοτήσεις. Και αυτό δυστυχώς το Συμβούλιο το έβαλε πάρα πολύ ωραία σε μια όμορφη ρήτρα που δεν μπορεί φαίνεται. Στο 72 το έβαλε το Συμβούλιο αυτό, στο συμβαστικό κείμενο. Θεωρώ λοιπόν ότι και αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη συζήτηση στα πλαίσια τραπεζικής εξυγίανσης, να κλείσουμε τέτοια πορτάκια παραθυράκια. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα η όλη διαδικασία εξυγίανσης, αν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Σας παρακαλώ λοιπόν να εργαστούμε γρήγορα, αποτελεσματικά, προκειμένου να έχουμε μια τραπεζική ένωση με ισχυρούς ευρωπαϊκούς ε, θεσμούς, όπως ζητούμε εδώ και τρία χρόνια από πλευράς του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σβέν, και τώρα εξ του ECR, των συντηρητικών, η κυρία Μπικηφόρ, σκιάδος συγγετριά. Σας ευχαριστώ. Ήταν ε, πραγματικά πολύ άξιο Έχω να επενέσω την προσέγγιση των πρασίνων που έχουν δύο εισηγητές. Ε, Δύο-τρία ζητήματα να αναφέρω. Καταρχάς, σκοπός όλης μας της δουλειάς σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό είναι να αποφύγουμε μεγάλες απώλειες και ζημίες και για τους καταθέτες και για τους επενδυτές και για το φορολογούμενο, αλλά να ελαχιστοποιήσουμε και τον κίνδυνο ε, επιμόλυνσης, αν θέλετε. Γιατί αυτό που μάθαμε από την κρίση είναι ότι η αβεβαιότητα προωθεί αλλά και δημιουργεί μια τέτοια διασπορά του κινδύνου. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να περιορίσουμε τον κίνδυνο και να υπάρχει ένα σωστό πλαίσιο εξυγίανσης. Συμφωνώ απόλυτα με όλους τους συναδέλφους που θεωρούν ότι αυτό είναι ο απότερος στόχος μας. Ωστόσο, τη γνωρίζουμε ότι ποτέ δεν είναι ίδια τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε ό,τι αφορά τις απώλειες και τις ζημίες των τραπεζών, γιατί αλλιώς θα μπορούσαμε να τα προβλέψουμε και να τα επιλύσουμε όλα εκ των προτέρων. Λοιπόν, καταρχάς, σε ό,τι αφορά την ευελιξία που χρειάζεται στην αντίδραση, αλλά και σε ό,τι αφορά την ε, δημοκρατική ευθύνη και λογοδοσία εκείνων που έχουν την εξουσία και την ευελιξία. Γιατί όποια και αν είναι αυτή η αρχή εξυγίανσης, θα χρειαστεί τελικά διάφορα εργαλεία, αλλά και αξιοπιστία και ευθύνη προκειμένου να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όταν χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά θα μπορούμε να τους ζητήσουμε απόδοση ευθυνών, να μας εξηγήσουν. Και αυτό που μας δίδαξε η Κύπρος είναι ότι οι αποφάσεις που ενδεχομένως επηρεάζονται από την Κομισιόν δεν, ε, τους, δεν τις ελέγχουμε δημοκρατικά τόσο πολύ όσο άλλες αποφάσεις. Θεωρούμε ότι αν ο Επίτροπος έχει πάρει μια απόφαση που ενδεχομένως να θέτουμε ένα αμφισβητήσει είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουμε αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να ζητήσουμε λογοδοσία για αποφάσεις επιτρόπων. Και παρόλα αυτά, δίνουμε στην Επιτροπή και στους Επιτρόπους τεράστια ε, εξουσία και σπανίως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα εργαλεία. Αν λοιπόν δώσουμε τέτοια εξουσία και αρμοδιότητα στην ε, Κομισιόν, θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ το θέμα της δημοκρατικής ευθύνης λογοδοσίας. Είτε στο σώμα των επιτρόπων, είτε και για τους μεμονωμένους επιτρόπους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της ευθύνη. για να υπάρχει αξιοπιστία σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων, θα πρέπει απαραίτητο να υπάρχει και ευθύνη σε ό,τι αφορά την αρχή εξυγίανση. Άλλο τώρα θα τι ισχύει για το ταμείο. Τι γίνεται όμως αν υπάρξει πτώχευση μιας μεγάλες ε, τράπεζης και ε, προκύψει ότι υπήρξε υπερβολική, υπερβολικό κούρεμα σε ό,τι αφορά τις απώλειες των ε, καταφετών. Ποιον τελικά θα καταγγείλουμε, ποιος θα είναι ο υπεύθυνος, η Επιτροπή, δεν υπάρχει μια κεντρική τράπεζα πίσω από αυτό. Πού είναι το backstop, πού είναι ο ανασταλτικό, προστατευτικός μηχανισμός σε αυτή την περίπτωση, σε περίπτωση που δεν είναι σωστή η απόφαση που ελήφθη. Ποιο τελικά είναι υπεύθυνο, αυτό είναι το ερώτημα που θέτω, σε ό,τι αφορά θέματα χρηματοδότηση. Κατανοώ γιατί κάποιοι λένε ότι θέλουμε να υπάρχει ένα κεντρικό ταμείο. Και καταλαβαίνω γιατί άλλοι πολιτικοί λένε ότι δεν έχουν ακόμα φτάσει στο σημείο αυτό που πραγματικά επιθυμούν κεντρικό ταμείο. Αν υπάρχει όμως ένα κεντρικό τέτοιο ταμείο, ένα δίκτυο τέτοιων ταμείων, δεν συμφωνώ με αυτά που μας λένε οι υπάλληλοι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν θα υπάρξει ποτέ χρηματοοικονομικός αντίκτυπος σε ό,τι αφορά την χρήση του ταμείου αυτού. Στην αρχή, όταν, όταν αρχίσαμε να εξετάσουμε την ενιαία επαπτική αρχή, τι λέγαμε, ότι αυτός που λαμβάνει, αυτός που τελικά πληρώνει το λογαριασμό, θα πρέπει να μπορεί να πάρει και την απόφαση. Ε, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος χρηματοοικονομικός αντίκτυπος. Οι χώρε που εμπλέκονται θα πρέπει να μπορούν να έχουν και λέγει κατά τη λήψη της απόφασης. αν κάποιο επιβάλλει κάποιο τέλος σε μια τράπεζα, θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια που ισχύουν όταν επιβάλλεται κάποιο τέλος σε κάποιο φορολογούμενο, σε κάποιο άτομο. Θα πρέπει αυτός που λαμβάνει την απόφαση, που πληρώνει, να μπορεί να λάβει και απόφαση. Αν η Κομισιόν τώρα υποστηρίξει ότι αυτό α, δεν θα πρέπει να θεωρείται, ε, δεν θα πρέπει να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων ο εμπλεκόμενος. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν θα το θεωρούμε εξορισμού κρατική επιδότηση. Νομίζω ότι θα ανακύψουν πολλά δύσκολα ερωτήματα. Τέταρτο σημείο. Δεν θα σας προκαλέσει έκπληξη. Υπάρχει ανησυχία σε ό,τι αφορά τον ρόλο των τρίτων χωρών και των μη συμμετεχόντων ε, κρατών μελών. Επαναλαμβάνω πράγματα που έχω πει και στο παρελθόν, αλλά στο SRM έχουμε δώσει στην ΕΙΜΑ μία δεσμευτική ε, λειτουργία διαμεσολόβηση σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία μεταξύ δύο αρχών διαμεσ... Ε, Αν στον ενιαίο μηχανισμό υπάρχει διαφορά απόψεων με μία αρχή εξυγίανση που δεν συμμετέχει η ΕΜΠΑ θα μπορεί να πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα πρέπει να κάνει και θα μπορεί νομικά ή πολιτικά να δώσει εντολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα δράσει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, γιατί μιλάμε για τεράστια ποσά χρηματικά. Αυτό θα πρέπει να το πετύχουμε σωστά. Να σκεφτούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτή η σχέση σε ό,τι αφορά αυτές τις δεσμευτικές απόψεις που θα λαμβάνονται. Αυτό ήταν το τέταρτο σημείο που ήθελα να αναφέρω. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Σύμφωνο απόλυτα με το Σβέν που αναφέρθηκε στην έλλειψη, ε, αν θέλετε, πεδίου ίσων όρων με, τις, ε, με τα ταμιευτήρια. Γιατί να παίρνουν αυτές ε, οι τράπεζες επιδοτήσεις. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας τομέας του τραπεζικού κλάδου που θα μπορεί να πει ότι σε διαρκή βάση μπορεί να απολαμβάνει διαφορετικούς όρους σε ό,τι αφορά τις εγγυήσει. Να μπορούν να δηλώνουν δηλαδή ότι δεν χρειάζονται να συμμετέχουν ανάλογα σε ό,τι αφορά τα τέλη προς το ταμείο αυτό. Δεν μπορούν να υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Να δούμε λοιπόν ποιες εξαιρέσεις έχουν δοθεί στον τομέα αυτών. Είναι ίσοι όροι, είναι δίκαιοι όροι. Δεν είμαι σίγουρη σε ό,τι αφορά δηλαδή τα δημόσια ταμιευτήρια, τους συνεταιρισμούς και τις ε, τράπεζε. τράπεζες. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα δημορφωθούν αυτοί οι όροι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Φόρτ. Ζήτησαν το λόγο η κυρία Χίνερ, Λάβενσον, Χόκμαρκ, Φλίν, Σάιμον, Πινκ, Φέιο, κυρία Ποδηματά και ο κύριος Λάμπερτς. Αλλά σε 40 λεπτά θα πρέπει να ψηφίσουμε. Γι' αυτό και δεν μπορώ να δώσω παραπάνω από 3 λεπτά στον κάθε ομιλητή. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν, να δώσω το λόγο στην κυρία Χιούνε. Χιούμπερτ, συγγνώμη. Ντανούτα. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι η πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπής είναι πολύ επικοδομητική και μας οδηγεί προς την ε, σύσταση των ε, θεσμών και των αρχών που λείπουν στο τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη. Γι' αυτό και χαιρόμαστε για τη θετική και επικοδομητική προσέγγιση και θα έχουμε και εμείς αντίστοιχη Άλλωστε, στόχος είναι η αποσύνδεση ε, των τραπεζών από τα δημόσια χρέη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ενιαίο μηχανισμό εξυγένσης και τις ε, τη σχέση του Συμβουλίου εξυγένσης και τι γίνεται με, τις, ε, με την οδηγία της ανάκαμψης εξυγένσης. Το Συμβούλιο Εξηγήσει ε, έχει μεγάλες αρμοδιότητες, αλλά δεν είναι σαφή η σχέση μεταξύ τη οδηγίας για την ανάκαμψη και εξυγίαση των τραπεζών και του SRM, του ενιαίου μηχανισμού εξυγίασης. Γιατί χρειάζονται από την οδηγία κατάλληλα σχέδια εξυγίασης, ενώ στο άρθρο 7 ζητήθηκε παραπομπή στην οδηγή για την ανάκαμψη και την εξυγίαση για να αποφευθεί επικάλυψη με τα υπάρχοντα σχέδια εξυγίασης. Μία λύση ίσως θα ήταν το Συμβούλιο Εξυγίασης να μπορεί να αναθεωρεί τα σχέδια που έχουν εκπονηθεί δυνάμει της οδηγίας ανάκαμψης και εξυγίασης των τραπεζών αντί να χρειαστεί από την αρχή να καταρτήσει ε, σχέδια. Σε ό,τι αφορά την τα δικαιώματα ψήφου στο Συμβούλιο εξηγήσει, πολύ σημαντικό θέμα, θέλουμε το σύστημα να είναι όσο πιο περιεκτικό γίνεται, να μην αποκλείει και ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας των αποφάσεων, πώς κατανέμε τα δικαιώματα ψήφου, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Και κοιτάζοντα όλα αυτά βλέπουμε ε, ότι τα κράτη-μέλη με ε, απλώς υποκαταστήματα και θηγατρικές ε, θα διτρέξουν τον κίνδυνο να έχουν ελάχιστα δικαιώματα ψηφοφορίας και να χάνουν στις ψηφοφορίες. Θα πρέπει να δούμε δύο εναλλακτικέ λύσεις. Αν θέλουμε να κρατήσουμε τη διαδικασία λήψη αποφάσεων όπως προτείνεται στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τότε τα κράτη-μέλη που έχουν υποκαταστήματα και θηγατρικέ θα πρέπει και αυτά τα κράτη να μπορούν να υποβάλουν ε, ε, σχέδια εξυγίασης πέραν αυτών που προτείνει το Συμβούλιο Εξυγίασης για κάθε περίπτωση. Ιδιαίτερα όταν διακυβεύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε ένα κράτος. Επίσης, μια άλλη εναλλακτική θα ήταν να δώσουμε στα υποκαταστήματα και στις θηγατρικές αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ανάλογα με αυτά που ε, ανταποκρίνονται στο μερίδιό τους ε, στην στον τραπεζικό κλάδο και στο πώς επηρεάζουν την αγορά. Και τέλος, για το πεδίο εφαρμογή του ενιαίου μηχανισμού εξυγίασης σε σχέση με τον ενιαίο υποπτικό μηχανισμό, γιατί με βάση τον ενιαίο υποπτικό μηχανισμό ε, θα είναι στενότερο το πεδίο εφαρμογή. Όλες οι μικρές τράπεζες θα εξακολουθούν να υπάγονται στις εθνικές αρχές εποπτείας. Οπότε όλες οι τράπεζες, άσχετες με το μέγεθός τους, ε, υπόκειται, στον ενιαίο μηχανισμό εξυγίασης. Θα υπάρχει πρόβλημα συντονισμού, αν η υποπτία γίνεται τοπικά, αλλά η εξυγίαση γίνεται κεντρικά. Θα πρέπει και αυτό το θέμα να το δούμε στον κανονισμό για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίασης. Ευχαριστούμε κυρία Χιούμπνερ, εκ μέρους των Σοσιαλιστών, το λόγο κύριο Σιαλούμπιστον. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπάρχει νομίζω ένα σημείο το οποίο αποδυναμώνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι ε, όσον αφορά την σύνθεση και, τον εκπροσώ, και τους εκπροσώπους του Συμβουλίου Εξυγένσης θα πρέπει ε, για το σημείο αυτό να προβλέψουμε πιο προσεκτικές διατάξεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι τους να γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει κάθε φορά που μία τράπεζα υπάγεται σε ένα σύστημα εξυγίανσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να συνεχίσουν να καταβάλλονται οι πληρωμές τους, να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις αποδοχές τους, ακόμα και όταν η τράπεζα βρίσκεται σε μια φάση εξυγίανσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης ε, η τράπεζα στη φάση αυτή να μπορεί να ενημερώνει τακτικά τους εργαζομένους και ο μηχανισμός εξυγένσης θα πρέπει να προβλέπει επίσης μια συγκεκριμένη ε, ένα συγκεκριμένο σύστημα ευθύνη και ενημέρωση, προκειμένου να, υπάρχει ένα σύστημα διαβούλευση με του εργαζομένου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι να αποτελούν ε, περιουσιακό και αυτή στοιχείο τη τράπεζα, ε, ένα σημαντικό κεφάλαιο τη τράπεζα και όχι απλώ ένα τμήμα τη τράπεζα το οποίο πλήττεται κάθε φορά που η τράπεζα αντιμετωπίζει προβλήματα. Εκ μέρους των φιλελευθέρων ο κύριος Κλίντς έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν βλέπουμε την κατάσταση των τραπεζών στις Ηνωμένες Πολιτείε, και αλλού βλέπουμε ότι είτε με αγορές είτε με συγχωνεύσεις οι μεγάλες τράπεζες ισχυροποιούνται ενώ οι μικρές οδηγούνται σε εξυγίαση. Γι' αυτό και το σύστημα χρειάζεται μία ενίσχυση γιατί είναι αρκετά εύθραυστο και ευάλωτο. Γι' αυτό και η πρόταση της κυρίας Φερέρ είναι πολύ σημαντική. Χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό εξυγίανσης, ιδιαίτερα για τις τράπεζες που έχουν διασυνοριακές δραστηριότητες. Βέβαια, στην πρόταση μιλάτε για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γιατί καλό είναι ε, να ισχύει για τις τράπεζες με διασυνοριακές δραστηριότητες, αλλά να έχουμε για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να δούμε και τις δραστηριότητες της ΕΚΤ. Και να δούμε αν μια τράπεζα ή μια χώρα συμμετέχει στην Ευρωζώνη ή όχι. Δεν θεωρώ ότι με το σύστημα προτείνεται θα καταλήξουμε σε καλά αποτελέσματα. Θα έχουμε δυσκολίες για να γεφυρώσουμε τα διαφορετικά συμφέροντα και θα τελικά θα τσακωθούμε για την χρηματοδότηση των ε, μεμονωμένων ε, φορέων. Δυστυχώς έτσι θα γίνει. Έτσι όπως ε, έχει γίνει η πρόταση θα καταλήξουμε σε πλήρη μη ικανοποίηση όλων των φορέων ποιοι έχουν τελικά ε, δικαίωμα ρύθμισης. Νομίζω ότι έτσι πραγματικά θα έχουμε προβλήματα και σε πολλές περιπτώσεις θα υπάρξει αδικία πραγματικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι χρειάζεται σε κάθε περίπτωση μία καλή εναρμόνιση των καθεστώτων εξυγίανσης, των εθνικών και των εθνικών ε, μηχανισμών ε, χρηματοδότησης. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα πετύχουμε αυτά έτσι γρήγορα και γι' αυτό θα απογοητευτούμε. Έχουμε φυσικά τις καλύτερες προθέσεις, αλλά δεν πρόκειται να τα πετύχουμε όλα αυτά. Μην ανησυχείτε. Έχετε έξι λεπτά μαζί με την υπόλοιπο χρόνο. Δυστυχώς αυτό είναι μεγάλο μειονέκτημα και νομίζω ότι η χρηματοδότηση θα μας προκαλέσει μεγάλα προβλήματα γιατί είναι σαφέστατο ότι εδώ και παραπάνω από 10 χρόνια το ταμείο αυτό δεν έχει τη χρηματοδότηση που θα έπρεπε να έχει και για το κατά πόσον οι ενδιάμεσες ε, λύσεις για μια πιστοτική γραμμή ή για χρηματοδότηση με άλλους ε, τρόπους. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι εφικτά όλα αυτά. Δεν ξέρω γιατί δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταμείο στο οποίο συμμετέχει κατά 27% ο Γερμανός φορολογούμενος για πράγματα και για που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με τη Γερμανία. Αυτό δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε στους πολίτες. Θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Κάτι άλλο τώρα για την διαθεσμική ασφάλεια. Σβέν, κάτι κατάλαβες λάθος. Αυτό που λέει ο Σβέν είναι το εξής. Δεν θέλει να εξαιρεθούν τα ταμιευτέρια, όχι. Θέλει ο Σβέν να κατοχυρωθούν αυτά στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν καταλάβατε καλά, συνάδελφε, τι είπε ο Σβέν. Και σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Αν τα εντρήματα αυτά αλληλασφαλιστούν και ε, φέρουν και οικονομική ευθύνη για την ασφάλιση αυτή, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μία λύση. Αυτό που θεωρώ, Σβέν, είναι ότι τα ταμιευτήρια θα πρέπει να επιλύσουν το πρόβλημα αυτό με διαφορετικό τρόπο. Ποιο συμμετέχει και ποιο όχι. Δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν ε, σε ένα σύστημα, αλλά όταν πρόκειται για εθνικέ τράπεζε να βγάζουν τον του απ' έξω και να τα ρίχνουν όλα στο φορολογούμενο. Αυτό όχι, δεν γίνεται. Κάτι τελευταίο τώρα. Ελπίζω να καταφέρουμε σχετικά γρήγορα να αποφασίσουμε σχετικά με τις ε, νομικές αυτές αμφιβολίες που υπάρχουν και να τις παραμερίσουμε γιατί δεν είναι δυνατόν να αποφασίζουμε για κάτι και τελικά εκ των υστέρων να προβάλλονται αυτές οι αμφιβολίες. Ευχαριστούμε κύριε Κλίντς. Ο κύριος Πίτερ Σάιμον για τρία λεπτά από τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και αγαπητέ Βόλφ για αυτό που είπες για τις δικαιολογίε που προβάλλονται σε ό,τι αφορά τα νομικά επιχειρήματα. Αλλά από τα Βερολίνα ακούμε το αντίθετο. Η Ευρώπη και ο φορολογούμενος ε, δεν απειλείται από τον τραπεζικό κλάδο, αλλά από τη γερμανική κυβέρνηση, γιατί μπλοκάρει τα πάντα η γερμανική κυβέρνηση αυτά. Τα αποφάσεις ε, της ΕΚΤ απορρίπτει και αρνείται την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξυγίανσης, τη χρηματοδότηση της εξυγίανσης, μα αν τα αρνούμαστε όλα αυτά, δεν προχωράμε ούτε ρούπι. Και ένα πράγμα μας βρίσκει σύμφωνος, ότι δεν θα πρέπει να, ε, να μην επιβαρυνθεί στο μέλλον ο φορολογούμενος. Και τι θα κάνει ο κύριο Σόιμπλε για να βγει από το φαύλο κύκλο. Ας έρθει και κάτι επικοδομητικό και θετικό πλέον από το Βερολίνο. Και εμείς θέλουμε όλοι να βρούμε το σωστό δρόμο για το μέλλον, αλλά δεν τα αρνούμαστε όλα και όλους. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο ελπίζω επιτέλους να φτάσει στο Βερολίνο πριν την επόμενη Κυριακή, προκειμένου κάτι επικοδομητικό να προτείνουμε πια ως λύση. Σας ευχαριστούμε κύριε Σάιμον. Το λόγο έχει ο κύριος Έπινγκ. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Πάντα με διασκεδάζει. Πάντα λέω με διασκεδάζει να ακούω τους Γερμανούς να μιλάνε για νομικά επιχειρήματα. Να σας θυμίσω ότι ο Μάρτιν Λούθερ κάποτε είχε πει ότι οι νομικοί είναι χριστιανοί. Ε, δεν ξέρω σε ποιους θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους νομικούς ή στις υπηρεσίες μας. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε υπέρ της εποπτείας του τραπεζικού συστήματος και είμαι και υπέρ του συστήματος εξυγίανσης επειδή θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πτώχευσης των τραπεζών και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και χρηματοδότηση. Πότε όμως θα, γεμ... πώς θα γεμίσει, πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό το ταμείο. Κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχουν δύο φάσεις ε, ε, στο τραπεζικό σύστημα. Ε, εποπτεία, εξυγίανση και κάποιοι άλλοι τρία βήματα ε, εποπτεία, εξυγίανση και το ευρωπαϊκό σύστημα ε, καταθέσεων. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν αυτό που αναφέρει ο κύριος Κλίντς είναι ακριβώς αυτό το σύστημα ε, αποταμίευσης κατάθεσης. Ο, η συγκεντρία θέλει ίσως εκεί να καταλήξει σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγυήσεων γιατί φυσικά ένα ταμείο ενδεχομένως να μην είναι γεμάτο. Μιλάμε για γραμμή πιστώσεων. Πώς ε, χρηματοδοτούνται αυτές οι γραμμές πιστώσεων σε ό,τι αφορά τον Ευρω... το γερμανό φορολογούμενο. Αυτά που έκανε τελικά ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Εξυγίανσης δεν είχε την αρμοδιότητα να διασώσει τις ε, τράπεζες και τελικά έγιναν όλα αυτά μέσω του Ισπανικού κράτους. χρησιμοποιήθηκε τελικά το ESM. Χτες ο Επιτρόπος Μπαρνιέ μίλησε για ένα public backstop, αυτούς τους ανθαλτικούς μηχανισμές. Αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησεων δεν χρησιμοποιείται ως όρος, αλλά έχω την αίσθηση ότι προς τα εκεί οδεύουμε. Αυτό με ανησυχεί, γιατί ένα τέτοιο σύστημα θα φροντίσει ε, να παίρνουν πιο, μεγάλους, ε, πιο μεγάλα ρίσκα οι μεγάλες τράπεζες, γιατί ξέρουν ότι θα υπάρχει κάποια τελικά δυνατότητα διάσωσης. Και αυτό αποτελεί ένα μεγάλο εθνικό ερωτηματικό εισηγήτρια. Να σας ρωτήσω τελικά μέσω του συστήματος που προτείνετε προς τα εκεί προς ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγυήσεων. Σας ευχαριστούμε κύριε Έπινγκ. Ο κύριος Φέιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι η έκθεση Φεραίρα ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση γιατί θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη σταθερότητα στο τραπεζικό σύστημα. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό. με, ιδιαίτερα μετά από τη διαχείριση που έγινε στο κυπριακό θέμα. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή χρήζει ιδιαίτερη προσοχή. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερα το θέμα τη διοίκηση του Συμβούλου Εξηγήσει και το σύστημα κατανομής των ψήφων. Σίγουρα θα χρειαστούν κάποιε τροποποίησεις εκεί που θα υποβληθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Σύμβουλο Εξυγίασης. Δεύτερον, το ίδιο το Ταμείο της Εξυγίασης χρήζει κάποιες ε, εμβάθυνσης ε, γιατί θα δημιουργηθεί μέσα σε μια δεκαετία με συνεισφορά των τραπεζών, πολύ σωστά όλα αυτά αλλά τι θα γίνει αν μέσα σε αυτή τη δεκαετία ανακύψει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και η λύση που θα βρούμε πρέπει να μας καλύψει για μετά τη δεκαετία, αλλά θα πρέπει να μας καλύψει και για το διάμεσο διάστημα. Γιατί θα είναι αργός ο ρυθμός σύστασης του Ταμείου εξηγήνσης από ό,τι φαίνεται. Θα ήθελα να το σκεφτεί λοιπόν αυτό η συγγετρία. Θα πρέπει να βρούμε μία λύση κοινοτική για να επιλύσουμε ενδεχόμενα προβλήματα που θα ανακύψουν στη διάρκεια της δεκαετίας, πριν την πλήρη λειτουργία του Ταμείου. Επίσης, ε, φαίνεται ότι η έκθεση αυτή ακολουθεί την γραμμή και τη έκθεσης Όκμαρ. Χόκμαρ. Λαμβάνοντας υπόψη τους καταθέτες. Θα πρέπει με την έκθεση αυτή να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους. Είναι σημαντικό να βγάλουμε τους καταθέτες από την εξηγήση των τραπεζών, αλλά θα πρέπει να δούμε με ποιους τρόπους θα προασπίσουμε την εμπιστοσύνη των καταθετών σε όλο το σύστημα. Αυτό είναι ένα σύστημα πολύ σημαντικό για την Τραπεζική Ένωση. Και σίγουρα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας το συμφέρον των καταθετών, είναι πολύ σημαντική η θέση τους και να ε, αποτρέψουμε οποιαδήποτε διαφυγή των καταθετών ε, θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των καταθετών και είμαστε πρόθυμοι να βρούμε λύσεις ε, στα πλαίσια της έκθεσης ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η θέση των καταθετών. Ευχαριστώ. Ε, Diego... Ευχαριστώ, Διέγκο. Το λόγο έχει η κυρία Ποδηματά τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και την ε, Ελίζα, την εισηγήτριά μας, για την αφοσίωσή της ε, και για την ε, προσέγγιση της σε ένα εξαιρετικής ε, σημασίας νομοθέτημα. Συμφωνούμε όλοι νομίζω ότι η δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης, το πακέτο της δημιουργίας της Τραπεζικής Ένωσης είναι ίσως η σημαντικότερη θεσμική παρέμβαση από συστάσεως της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης είναι η πιο σημαντική, είναι εξίσου σημαντική θεσμική παρέμβαση με την ίδια την απόφαση δημιουργίας του ευρώ. Ψηφίσαμε ήδη στο Στρασβούργο τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας και όπως τόνισε και η Ελίζα στην εισήγησή της, αλλά και ο Επίτροπος Μπαρνιέ χθε, η ενιαία αρχή εκαθάρισης τραπεζών και το ενιαίο κοινό ταμείο εκαθάρισης τραπεζών είναι το επόμενο αναπόδραστο και αναπόσπαστο τμήμα για τη δημιουργία της τραπεζικής ένωσης. οι ενιαίοι κανόνες παντού και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία και σε ό,τι αφορά την εποπτεία και σε ό,τι αφορά την εξυγίανση και την εκαθάριση τραπεζών χωρίς τις τρευλώσεις που αναπόφευκτα δημιουργούνται όταν ο τελικός λόγος ανήκει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές αναφέρθηκαν διάφοροι συνάδελφοι στην πολύ ε, οδυνηρή και ακριβή για τους φορολογούμενους, τους Κύπριους φορολογούμενους, λύση που επιβλήθηκε στην Κύπρο. Ε, ο μόνος τρόπος λοιπόν, οι ενιαίοι κανόνες παντού είναι ο μόνος τρόπος για να υπερβούμε τον κατακαιρματισμό, να, μειώσουμε, να περιορίσουμε τους κινδύνους, να μειώσουμε τις ανισότητες μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ανάμεσα στο βορρά και το νότο και να τα αποσυνδέσουμε από το ρίσκο της χώρας που όπως ξέρουμε ακόμα και σήμερα αυτό το ρίσκο της χώρας δημιουργεί πιστωτική ασφυξία στις χώρες που κυρίως χρειάζονται ρευστότητα και υπερβολικά σχεδόν απαγορευτικά επιτόκια δανεισμού για τις επιχειρήσεις κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτών των χωρών. Ε, αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να τα υπερβούμε άμεσα για να βοηθήσουμε τη συνολική ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας και την συνολική ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. θέλω ένα σημείο να επισημάνω και να ενώσω τη φωνή μου με αυτήν του συναδέλφου διέγκο ε, φέιο που μίλησε αμέσως πριν ε, από μένα. χαίρομαι καταρχήν που οι βασικές τοποθετήσεις των σκιωδών και όλων μας κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση το σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι ε, ο τραπεζικός τομέας θα παραμένει κατακαιρματισμένος και ευάλωτος όσο καθυστερεί η εφαρμογή αυτού του νέου πλαισίου και ξέρουμε πολύ καλά ότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι να τεθεί ε, πλήρως σε λειτουργία αυτό το πλαίσιο. Θεωρώ λοιπόν και εγώ ε, ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την πιθανότητα να εισάγουμε σε αυτόν τον κανονισμό κάποιες μεταβατικές διατάξεις κάποια μεταβατικά μέτρα μέχρι δηλαδή να συσταθεί και να αποκτήσει δύναμη πυρός το ταμείο ε, εκαθάρισης ε, και αυτό που σκέφτομαι ε, αλλά μπορούμε να εξετάσουμε διάφορες εναλλακτικές η ιδέα που σκέφτομαι είναι να μπορεί να παίξει μεταβατικά μέχρι να συσταθεί και να λειτουργήσει αυτό το ενιαίο ταμείο εκαθάρισης να μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο ο esm ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας που άλλωστε έχει συνδεθεί και με την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ασφαλώς με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. νομίζω ότι είναι σημαντικό να επιδιωχθεί μια τέτοια συμφωνία για τη μεταβατική περίοδο πριν από τα stress test από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γιατί ε, τυχόν αρνητικά αποτελέσματα σε αυτά τα stress test, τα τεστ αντοχής μπορεί να οξύνουν την τραπεζική αλλά και τη δημοσιονομική κρίση εάν δεν είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι να τα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε Εκ uh, Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ την εισηγητριά μας για την παρουσίαση που έκανε, καθώς επίσης και τους άλλους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Μία πρώτη παρατήρηση θέλω να κάνω. Πραγματικά πρέπει να τονίσω αυτό το οποίο είπε η κυρία Φερέιρα, ότι όντως το σύστημα αυτό θα πρέπει να συνάδει με την οδηγία για την ανάκαμψη και την εκαθάριση, την εξυγίανση. Και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος κανόνας θα εφαρμόζεται κάθε φορά. Δεύτερη τώρα παρατήρηση. Μια σκέψη που θέλω να κάνω σε σχέση με τη συζήτηση που είχαμε. Ξέρω ότι μερικέ φορέ συζητάμε για το χρηματοπιστωτικό τομέα σαν να μην έχει καμία σχέση με την οικονομία, με τη γενική οικονομία. Και αυτό όμω δεν ισχύει. Ο χρηματοπιστωτικό τομέα δεν είναι μια ξεχωριστή οντότητα, αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα τη οικονομία και η κρίση την οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει να κάνει με προβλήματα τη πραγματική οικονομία. Έχουμε ύφεση, έχουμε τιμέ οι οποίε καταραίουν, όλα αυτά συνδέονται με το χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίο πολλέ φορέ δεν κάνει σωστά τη δουλειά του και πολλέ φορέ επιδεινώνεται τελικά. Θεωρώ πάντω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια σφαιρική εικόνα των πραγμάτων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε το ακόλουθο. Κάθε φορά που έχουμε μια συστημική κρίση, ξέρω ότι μερικές φορές ε, συζητάμε τις κρίσεις εντελώς μονομένα. Οι τραπεζικές κρίσεις μόνες τους, για παράδειγμα. Κάθε φορά που υπάρχει μια συστημική κρίση, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το σύνολο της οικονομίας... βρίσκεται σε πολύ δινή θέση. Και τότε ακριβώς θα πρέπει να εξασφαλίζουμε όχι μόνο ότι έχουμε αποφάσει εκαθάριση σωστέ, αλλά ότι, λαμβάνουμε τις απαραίτητες, ότι έχουμε τις απαραίτητες ικανότητες εκαθάρισης. Και συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην βρισκόμαστε σε καταστάσεις τέτοιες όπου έχουμε κυβερνήσεις, αρχές ε, και ούτω καθεξής που θεωρούν ότι άλλοι τελικά είναι υπεύθυνοι για την επίλυση των προβλημάτων. Κάθε φορά που έχουμε μια μεγάλη συστημική κρίση θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ακόμα και ένα μεγάλο Ευρωπαϊκό Ταμείο Καθάρισης δεν θα είναι ποτέ σε θέση και δεν θα αρκεί από μόνο του για να επιλύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Και τότε ελοχεύει ο κίνδυνος της μετάθεσης του προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να νομίζουμε δηλαδή ότι αυτό από μόνο του επιλύει το ζήτημα. Πρέπει να γνωρίζουμε επίση και ποια είναι τα χρήματα τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ ότι σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή συστημική κρίση τα χρήματα αυτά δεν πρόκειται να φτάσουν. Γι' αυτόν τον λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια νομική σαφήνεια και διάκριση για κάθε κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε, για όλα τα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ξέρετε ότι ε, η λειτουργική επιχειρησιακή σαφήνεια απαιτεί και νομική σαφήνεια. Και ελοχεύει ο κίνδυνος τελικά να εγκρίνουμε τον, την νομοθεσία αυτή, προτού τελικά καταφέρουμε να εγκρίνουμε την οδηγία για την ανάκαμψη και την εκαθάριση. Και θεωρώ επίση ότι διατρέχουμε και τον κίνδυνο να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πάρα πολλές μεγάλες απαιτήσει από τον κανονισμό αυτό. Πρέπει αντίθετα να δούμε πώς τα πράγματα θα λειτουργήσουν στην πράξη, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρειαστεί να λάβει κάποιες αποφάσεις και όταν η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα πρέπει και αυτή με τη σειρά της να διαμεσολαβήσει. Ξέρετε ότι υπάγεται ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αρχή αυτή και δεν είναι ανώτερη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα δημιουργηθεί μια περίεργη κατάσταση και πολλές φορές μπορεί να υπάρχει και μια σύγχυση όσον αφορά τις αρμοδιότητες που φέρει ο κάθε φορέας. Θεωρώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σαφήνεια στο τι κάνουμε ακριβώς κάθε φορά που έχουμε μια μεγάλη τραπεζική κρίση. Ποια είναι η ευθύνη που φέρουν τα κράτη-μέλη και φέρουν τα κράτη-μέλη κάποια ευθύνη στην περίπτωση αυτή. Όταν έχουμε μια μεγάλη συστημική κρίση, πώς αντιμετωπίζουμε το γεγονός ότι θα υπάρχουν τελικά διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικές δομές και διαρθρώσεις εντός και εκτός Ευρωζώνης. Ενώ παράλληλα γνωρίζουμε όλοι ότι ο τραπεζικός μας τομέας είναι πλέον εντελώς διασυνοριακός. Πρέπει επίσης να πω κάτι ακόμα. Ελπίζουμε πραγματικά ότι θα πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα με το σύστημα εκαθάρισης αλλά φοβάμαι ότι έχουμε περισσότερο, νεότερο βαθμό ελπίδας και χαμηλότερο βαθμό αξιοπιστίας αυτή τη στιγμή. Αν δεν καταφέρουμε να αφησίσουμε περισσότερη αξιοπιστία στο κείμενο αυτό, τότε νομίζω θα αποτύχουμε. Γι' αυτό το λόγο απευθύνομαι προς την εισηγήτρια λέγοντας ότι χρειαζόμαστε απαραίτητη νομική σαφήνεια και δεν λέω ότι δεν έχουν κάποια αξία τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, τα νομικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και ότι μπορούμε από την μία νυχτή να τα διαγράψουμε. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ο απαραίτητο σεβασμός για τη νομική σαφήνεια την οποία χρειαζόμαστε στο κείμενο αυτό. Αν δεν υπάρχει νομική σαφήνεια στο κείμενο, δεν έχουμε και εξοπιστία. Σε ευχαριστώ, Πάμπλο. Δύο παρατηρήσεις όσον αφορά την σαφήνεια και την αξιοπιστία. Θα ήθελα να αφαιρθώ καταρχάς στο Ταμείο Καθάρισης. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να φέρουμε μία γραμμή διάκρισης ως προς τις αρμοδιότητες του Ταμείου αυτού. Γιατί ξέρετε ότι ε, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ανάμεσα στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με συγχωρείτε. Ξέρετε ότι πολλέ φορέ το Συμβούλιο προχωρά ακόμα και σε αρμοδιότητες ανακεφαλοποίηση τραπεζών και αυτό το διαφέρει πάρα πολύ από τη γραμμή την οποία ακολουθούμε εμεί. Νομίζω επίσης ότι το Ταμείο αυτό θα πρέπει να έχει μεγαλύτερες διαστάσεις. Αν το Ταμείο βέβαια πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, τότε ενδεχομένως να δοθούν λανθασμένα κίνητρα στις τράπεζες και να λάβουν πάρα πολύ ψηλό κίνδυνο γιατί θα γνωρίζουν τελικά ότι έχουν ένα συλλογικό συμφέρον, να θέλετε, κατά το ταμείο αυτού. Αν είναι πολύ μικρό όμω το ταμείο, τότε ουσιαστικά θα επιτελέσει μόνο γραφειοκρατικέ ε, διαδικασίε. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να βρούμε εμεί την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στο να έχει υπερβολικέ ή χαμηλέ αρμοδιότητε το ταμείο αυτό. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση που ε, θέλω να κάνω. Δεύτερη τώρα παρατήρηση. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ουσιαστικά αντιγράψει στο κείμενο εδώ την θέση του Συμβουλίου και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα φιλικό απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο κείμενο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού δεν κάναμε κάτι τέτοιο, δεν αντιγράψαμε σε καμία περίπτωση το CRD4. Για ποιο λόγο κάναμε κάτι τέτοιο όμως στο δικό μας το κείμενο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να υπάρχει επικάλυψη νομικών κειμένων όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Διαφορετικά δίνουμε την εντύπωση ότι ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για τα κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν στον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης, πράγμα το οποίο δεν πρέπει να ισχύει. Μία ακόμη παρατήρηση. Ξέρετε ότι ε, η αρχή εκαθάρισης ε, και όλες οι αρμόδιες αρχές ε, θα πρέπει να είναι σε θέση να δούνε ποιος είναι ο βαθμός φερεγγιότητας και ποιος είναι ο βαθμός καθάρισης των τραπεζικών συστημάτων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε ότι υπάρχουν δύο δυνατότητες. Είτε μπορούμε να ζητήσουμε από μία τράπεζα να αναθεωρήσει το σχέδιο το οποίο έχει αναδιάρθρωσης, αλλά στην περίπτωση αυτή, σε ορισμένε περιπτώσεις, δεν θα είμαστε σε θέση να επιλύσουμε ή να καθαρίσουμε μια συστημική τέτοια τράπεζα εξαιτία της κατάστασης που θα ισχύει ώστε θα καταφέρουμε ουσιαστικά να αποφύγουμε ότι η εκαθάριση, η εξυγίανση ενός τραπεζικού συστήματος, μιας τράπεζας, ενός ομίλου, δεν θα έχει στη συνέχεια δευτερογενείς επιπτώσεις στον υπόλοιπο τραπεζικό κλάδο. Όσον αφορά τώρα τον ενιομηχανισμό εξυγίανσης, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ότι στην περίπτωση που μια τράπεζα είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχει πάρα πολύ μεγάλες διασυνδέσεις και δεν μπορεί να καθαριστεί, τότε θα πρέπει να μειωθεί το μέγεθός της ή να μειωθεί ο βαθμός διασύνδεσής της προκειμένου να μπορεί να ενταχθεί στο σύστημα εκαθάρισης. Επίσης χρειάζεται ένας υψηλός βαθμός πειθαρχία στα πλαίσια των χωρών που θα συμμετέχουν στο σύστημα SRM, ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης. Τότε κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να επιλύσουμε ένα 80% των προβλημάτων. Να πω ακόμη ότι ε, το κείμενο αυτό και το κείμενο για την ανάκαμψη και την εξυγίαση των τραπεζών έχει να κάνει με την εξυγίανση συγκεκριμένων ε, πιστοτικών ιδρυμάτων. Όταν μιλάμε για όλο όμως τον κλάδο ή για την αντιμετώπιση συστημικών κρίσεων, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο αυτό το κείμενο για να λύσουμε μια συστημική κρίση. Σας ευχαριστούμε κύριε Λάμπερτς. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις σύντομες και να παρουσιάσω τις σκέψεις μου. Σίγουρα χρειαζόμαστε ασφάλεια δικαίου και νομική σαφήνεια, όπως ε, ανέφερα πολλοί συνάδελφοι, αλλά κάτι άλλο εξίσου σημαντικό είναι να τηρήσουμε τις ημερομηνίε εφαρμογής του δεύτερου πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης. Όπως είπε και χθε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Γερμανία, η εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης θα επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψη. Συμφωνώ απόλυτα λοιπόν με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, αυτή θα πρέπει να είναι και η δική μας προτεραιότητα και της Επιτροπής μας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιταχυνθεί η οικονομική ανάκαμψη. Ιδιαίτερα σε αυτή την συγκυρία που βρισκόμαστε. Το Κοινοβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή Ένεκρινε πολλές εκθέσεις, το Τούπακ, το διπλό πακέτο, το εξαπλό πακέτο, το, Εποπτεία. Έχουμε τώρα την τελευταία ευκαιρία, την τελευταία μεγάλη πρόκληση της παρούσας κοινοβουλευτικής θητείας και πιστεύω ότι ακριβώς επειδή είναι η τελευταία μεγάλη πρόκληση είναι κεφαλαιόδου σημασία να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Κύριε Φερέιρα, θέλετε να ακούσουμε ε, σύντομα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί αν δεν κάνω λάθος, αρκετοί συνάδελφοι περιμένουν τα σχόλια και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εκπρόσωπό της και στο τέλος στην εισηγητριά μας την κυρία Φερέιρα. Thank you. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την κυρία Φερέιρα και όλους ε, που έλαβαν το λόγο. Σας ευχαριστώ για τα επικοδομητικά σας σχόλια. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, η πρόταση αυτή είναι θεμελιωδού σημασία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρούμε ότι πρόκειται για τον τρίτο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης και αυτός ο πυλώνας θα πρέπει το των δυνατών να καταστεί λειτουργικό. Γι' αυτό λοιπόν ασκούμε μεγάλη πίεση προ το Συμβούλιο. Θεωρούμε ότι το Κοινοβούλιο και αυτό θα πιεστεί ιδιαίτερω προκειμένου να υποβάλει μια σωστή λύση για την πρόταση αυτή το συντομότερο δυνατόν. Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε τις συζητήσεις της Επιτροπής από πλευράς Κομισιών. Είναι βασικό σε αυτή την πρόταση να παραμείνουν τουλάχιστον όλες οι επιτυχίες που έχουν να κάνουν με την κεντρική διαμόρφωση του συστήματος. Μία ενιαία αρχή θέλουμε και θέλουμε και ένα ενιαίο ταμείο. Γιατί θεωρούμε ότι αυτός είναι ο πιο σωστός τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης. Επίσης, θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι η πρόταση αυτή βασίζεται στον BRD. Άρα, όλα τα βασικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με την συμμετοχή του προλογούμενου. με τη συμμετοχή του Ταμείου Εκαθάρισης σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό της εκαθάρισης, τη εξυγένση, όλα αυτά θα ρυθμίσονται στον BRD, που θα είναι Ε, σε ό,τι αφορά την ανάκαμψη για τι εξηγήσει των τραπεζών. όλα αυτά θα πρέπει να τα πούμε. Θα πρέπει να σα πω ότι συμφωνώ και με τον επικεφαλή της BRD. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε όλα όσα έχουν να κάνουν με το... Επίσης, θα πρέπει να συζητήσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με το χρηματοοικονομικό αντίκτυπο. Αναφέρθηκε αυτό. Ε, θέματα σε ό,τι αφορά τις τρίτες χώρες, σε ό,τι αφορά την συμμετοχή των ε, αρχών των υπηρεσιών ε, της χώρας υποδοχής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει μια επικοδομητική συζήτηση για όλα τα θέματα αυτά. Και τέλος πρέπει να πούμε ότι προσβλέπουμε και στην έκθεση της κυρίας Φρέιρα. Και παρακολουθούμε ασφαλώς τις συζητήσεις εδώ στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Φερέιρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Σημείωσα επιμελώς ε, τις ανησυχίες και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων και έχουμε πια πολύ υλικό για να βελτιώσουμε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ ε, επιβεβαίωσα την αρχική μου πεποίθηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ιδιαίτερα επικοδομητική στάση και ήδη έχουμε μία συμφωνία επί της αρχής για το νομικό πλαίσιο που προτείνει στην πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα απλώς να πω ότι προέκυψαν ορισμένα βασικά θέματα εργασίας ε, για τη σύντομη περίοδο που έχω να εκπονήσω την έκθεσή μου. Ένα από τα θέματα αυτά είναι, όπως είχα πει και εγώ στην αρχή, είναι το θέμα του εκτελεστικού διευθυντή του Συμβουλίου Εκαθάρισης, το θέμα της λογοδοσίας για τις αποφάσεις και η αποσαφήνιση των σχέσεων του Συμβουλίου Εκαθάρισης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και πολλοί συνάδελφοι επισήμαναν αυτά τα ζητήματα, τα επιμέρους. Ένα δεύτερο θέμα αφορά το κεντρικό άξονα του συστήματος και θα πρέπει μεταξύ μας να συνεννοηθούμε και να διευκρινίσουμε ότι η ενιαία υποπτία μας οδηγεί σε ενιαίο μηχανισμό εκαθάρισης και απαιτεί και ένα ενιαίο ταμείο εκαθάρισης. Και καλό θα ήταν να υπενθυμίσουμε ότι η λειτουργία αυτού του Ταμείου Εκαθάρισης, εκαθάρισης και Εξυγίασης δεν είναι να λειτουργήσει ως Ταμείο Διάσωσης. Ο ρόλος του Ταμείου Εκαθάρισης δεν είναι να υποκαταστήσει τους φορολογούμενους. Γιατί αυτό ουσιαστικά έκαναν οι φορολογούμενοι μέχρι τώρα, διάσωσαν τι τράπεζες. Αλλά το Ταμείο Εκαθάριση, οι εξηγήσεις, είναι ε, για να διευκολύνει του μηχανισμού ε, καθάρισης και όχι για να πληρώσει τα σπασμένα της εκαθάριση. Για γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το σύστημα του bail-in, τη διάσωσης με ίδια μέσα των τραπεζών δηλαδή. Οπότε, όταν πολλοί ευρωβουλευτές είπαν ότι θα πρέπει το Ταμείο από την αρχή να είναι ε, πρικοδοτημένα με πολλά κονδύλια και όταν μιλούμε για κάποιες δημοσιονομικές γραμμές θα πρέπει να το διορθώσουμε. Δεν θα πρέπει φορολογούμε ε, να χρηματοδοτήσουμε το ταμείο. Μπορούν μεν στην αρχή να έχουμε μια δημοσιονομική γραμμή, αλλά αυτή θα την ε, ε, πληρώνουν ουσιαστικά οι τράπεζε όταν αποκτήσει το σύστημα μεγαλύτερη σταθερότητα. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε του φορολογούμενου να διασώζουν τι τράπεζε και τώρα θα περάσουμε σε μια άλλη κατάσταση όπου οι ίδιοι οι μέτοχοι ή οι ιδιοκτήτε τη τράπεζα, ανάλογα με την ιεράρχηση του εστιάσου με τα ίδια μέσα, αυτοί θα πληρώνουν, ε, θα αναλαμβάνουν το κόστο ε, τη καθάριση τη πτώχευση. Απλώ θα διευκολύνεται η θέση σε λειτουργία αυτή τη διαδικασία από το ενιαίο ταμείο. Γι' αυτό μιλήσαμε για τη χρηματοδότηση να έχουμε διαθέσιμη μία ε, δημοσιονομική γραμμή για να μην είναι το Ταμείο ένας χάρτινος τίγρης όπως μας είπε ο Φίλιπ Λάμπερτς. Μόνο στα χαρτιά δηλαδή να φαίνεται. Τώρα σε ό,τι αφορά τα κριτήρια της ανακεφαλαιοποίησης ε, με βάση το μηχανισμό σταθερότητας αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να είναι γνωστά και να έχουν στενή σχέση με τη λειτουργία του συστήματος ολόκληρο. Γιατί αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι η ισορροπία της εσωτερικής αγοράς και ανάγκη εξασφάλισης της ε, αποφυγής διαστρέβλωσης αυτών των κοινών κανόνων μέσω κάποιων άλλων στοιχείων που δεν στηρίζονται στη διαφάνεια ή δεν είναι γνωστά από όλους. Οι κανόνες λοιπόν θα πρέπει να είναι σαφείς, διαφανείς και κοινοί, ενιαίοι. Τώρα, σε σχέση με τη θέση σε εφαρμογή του συστήματος. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και με το μηχανισμό μετάβασης. Το ταμείο θα πρέπει να είναι γερό, στεναρό και να δούμε πώς θα συνδυάσω αυτό το σύστημα με τα εθνικά συστήματα και με τα εθνικά ταμεία εκαθάρισης που υπάρχουν. Και το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό της διάρθρωσης. Ένα άλλο ζήτημα που προέκυψε από τη συζήτηση είναι η ανάγκη συνοχής του συστήματος. Η συνοχή αυτή θα πρέπει να φανεί στην, στον παραλληλισμό με την Οδηγή για την ανάκαμψη και την εξηγένση των τραπεζών, την BRRD. Θα πρέπει να συνδυάσω αυτά τα δύο κείμενα, για το πρώτο είναι ο εισηγητής ο κύριο Χόκμαρκ. Ο Φιλίπ Λάμπερτς είπε ότι το κείμενο που μας υποβλήθηκε για συζήτηση είναι το κείμενο του Συμβουλίου, κάτι που δημιούργησε προβλήματα σε ορισμένες περιπτώσεις. Εγώ είμαι σκιώδη συγγήτρια για την οδηγία για την ανάκαμψη και εξηγία των τραπεζών και θέλω στο μέτρο του δυνατού να συγκλίνουν τα δύο κείμενα, να μην είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Χρειάζεται η συνοχή και ένα εχέγγυο της συνοχής είναι αυτό που μας είπε η Σιλβί Γκουλάρ. Θα πρέπει να έχουμε μεταβατική και εύρυθμη μετάβαση μεταξύ του επόπτη και, του, και της αρχής ε, εξηγίασης. Θα πρέπει η μετάβαση αυτή να γίνει με εύρυθμο και ομαλό τρόπο. Επίσης, όπως είπε ο κύριος Σέγμαν, έχουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και κάποιων ε, στοιχείων που βρίσκονται εντός εκτός του συστήματος. Θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που είπαν κάποιοι συνάδελφοι και κυρίως ο κύριος Λούντβιχστον και που υπάρχει στην οδηγία για την ανάκαμψη, των και εξηγέση των τραπεζών την κοινωνική ευθύνη στη διαδικασία καθάρισης. Λαμβάνουμε υπόψη και αυτό το θέμα στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξηγέση των τραπεζών και επίσης είναι προφανές ότι είναι σημαντικό να έχουμε και στο σημείο αυτό μια ρήτρα αναθεώρησης. Τέλος, φιλοδοξούμε να εργαστούμε με ταχύς ρυθμούς. Αυτό βέβαια θα γίνει εις βάρος της ποιότητας του έργου μας. Γι' αυτό και ζητώ τη βοήθεια και υποστήριξη της γραμματείας στην προσπάθεια αυτή για να δούμε πού μας παίρνει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα χωρίς όμως να διακυβεύουμε την ποιότητα των εργασιών. Δεν μπορούμε να προτρέχουμε και πολύ του Συμβουλίου, γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί να το περιμένουμε. Πάντως, γνωρίζουμε ότι τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θυσιάσουμε την ποιότητα στο βωμό της ταχύτητας. Γιατί το χρονοδιάγραμμα ήδη είναι γνωστό και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι τα τέλη του έτους μια απόφαση. Εγώ θα τηρήσω το χρονοδιάγραμμα που έχει προβλεφθεί. Θα προσπαθήσουμε στο μέτρο του δυνατού να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Όχι όμως εις βάρος της ποιότητας. Γιατί, επαναλαμβάνω, υπάρχουν πολλά στοιχεία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ θερμότατα όλους τους ε, συναδέλφους για τη συνεργασία τους. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις τους. Και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το κεντρικό σημείο όλων αυτών, το βασικό στόχο Τη νομοθεσίας, που είναι μια εύρυθμη εσωτερική αγορά, ένα πιο πάγιο, σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα, ικανό να λειτουργεί και να στηρίζει την πραγματική οικονομία, προστασία των φορολογουμένων, ώστε να μην είναι αυτοί που θα πληρώνουν τις εκαθαρίσεις, αλλά οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των τραπεζών, οι μέτοχοι των τραπεζών ή ο ίδιος ο τραπεζικός κλάδος θα πρέπει να πληρώνει τις διαδικασίες εκαθάρισης, εξυγίασης και επίσης να εξασφαλίσουμε μια σταθερότητα για τους ε, πολίτες που θα πρέπει ε, να μπορούν ε, οι ήσυχοι να καταθέτουν τα χρήματά τους στις τράπεζες. Άλλωστε το FDIC έδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα όραμα προς το οποίο βαίνουμε και εμείς. Άλλωστε ο Βόλφ Klintz μας υπεθύμησε αυτό το θέμα και πολύ συχνά μας λέει ότι στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα για τους μεμονωμένους καταθέτες, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπονομεύεται από το νέο σύστημα διαχείρισης των τραπεζών. Σας ευχαριστώ θερμά αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμβολή της και ελπίζω ότι αυτό το πνεύμα συνεργασίας ε, θα φέρει σε αίσιο πέρα σε αυτές τις διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρώσουμε την κοινοβουλευτική μας θητεία με μια καλύτερη κατάσταση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Ευχαριστώ Ελίσσα η εξέταση της, του σχεδίου έκθεσης γίνει στις 14 Οκτωβρίου και η προθεσμία για τις τροπολογίες λήγει καταρχήν στις 18 Οκτωβρίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου και στην Ολομέλεια του Μαρτίου θα λάβει χώρα η τελική ψηφοφορία. Προχωρούμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημέρησης διάταξης, τις ανακοινώσεις. Σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και ΚΟΝ για την ε, νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της στις 12 Σεπτεμβρίου να εφαρμόσει το κανόνα 51, τη διαδικασία μεικτή αρμοδιότητας. Οπότε η γραμματεία της Επιτροπής ε, Πολιτικών Ελευθεριών και της δικής μας θα προτείνουν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα για τις κοινέ εκθέσεις, για την οδηγία ε, κατά το ξεπλήματος ε, ε, χρήματος και της μεταφοράς κονδυλίων. Θα ψηφίσουμε και για τις εκθέσεις εκθέσεις το αργότερο τον Ιανουάριο. Και ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ανάγνωση τρεχούσης της κοινοβουλευτικής θητείας εξέταση των τροπολογιών της έκθεσης ε, έχει προβλεφθεί, που είχε προβληθεί και σήμερα φυσικά αναβάλλεται. Τώρα, σήμερα το απόγευμα θα έχουμε συνάντηση με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων στα πλαίσια της συζήτησης των τροπολογιών της έκθεσης της ΕΚΟΝ για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο με εισηγήτρια την κυρία Φερέρα. Ε, το Συμβούλιο πριν τις, ε, πριν τις θερινές διακοπές είχε ε, εγκρίνει κάποια συμπεράσματα και στα πλαίσια των αποφάσεων που μπορούν να ληφθούν σε ένα κράτο μέρο και ίσω ε, έχουν επιπτώσει και σε άλλα κρατημέλη, έχει νόημα να συζητήσουμε το απόγευμα το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τον κύκλο του 2013. Τώρα θα πρέπει να εγκρίνουμε και το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεών μα για το επόμενο έτο. Έχετε λάβει στον ντοσέ σα τι προτάσει και ελπίζω να μην έχετε αντιρρήσει. Οπότε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ψηφοφορίες. Στο σημείο 10 τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα με εισηγήτρια την Περβάνς Μπερές έχει αναβληθεί για μεταγενέστερη ψηφοφορία οπότε θα ψηφίσουμε σήμερα την τελική συμβαστική λύση ε, για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέση με εκτελεστικό διοικητικό στελεχών των εισηγουμένων στο χρηματιστήριο εταιριών. Έκθεση Κράτσα και Ρέγνερ είναι αρμόδιες επί της ουσίας και η γνωμοδότηση είναι και από τη δική μας επιτροπή. Άρχεται η ψηφοφορία. Σβέν, έχεις ηλεκτρονική κάρτα μαζί σου. Όχι. Ούτε κυρία Μπέρες. Άρχεται η ψηφοφορία για δοκιμαστική καταρχήν ψηφοφορία. One more. No. Χρειάζεται κάποια δοκιμή. Όχι. Ναι, Ωραία. Συμβιβαστική α, υπέρ. Σβέν. Α, ναι, συγγνώμη, ο εισηγητής ζήτησε το λόγο. Κύριε Σμιθ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για ένα κείμενο πραγματικού συμβιβασμού, κοινοβουλευτικού συμβιβασμού. Ξεκίνησα στο ένα σημείο και τελείωσα σε ένα τελείω διαφορετικό σημείο. Βρίσκομαι εδώ και συμμετέχω στο κοινοβούλιο εδώ και πάρα πολύ καιρό και ξέρω ότι αν θέλουμε να πετύχουμε αποτελέσματα. Πραγματικά πρέπει να ακούμε και να συμβαζόμαστε, να ευχαριστήσω τους βοηθούς, τους φλευτές, τη γραμματεία όλος ιδιαίτερος. Ελπίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, σε τελική ανάλυση να μπορέσουμε να δώσουμε μία έκθεση. Ιδάλλως θα καθόμαστε εδώ σαν κότες και θα παρακολουθούμε αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο αμέτωχοι. Ακόμα και αν δεν μας αρέσουν όλα τα στοιχεία της έκθεσης, νομίζω ότι μπορούμε κάτι να πετύχουμε με αυτήν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σμιθ και πολύ λυπάμαι που ξέχασα να σας δώσω το λόγο. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Συμβαστική α. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική β. Υπέρ. Κατά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 Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Ηλεκτρονικά ελέγχουμε το τρίτο τμήμα. Ε, Ο Σβέν είναι κατά. Και άλλε δύο ψήφοι λοιπόν κατά. Πέρασε ψηφοφορία, εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα παρακαλώ. Τροπολογία του εισηγητή. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις θα ψηφίσουμε την τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά αν θέλετε το ελέγχουμε. Είσαστε κατά και Ιαν και ο Σβέν. So we close the vote. Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται. 22 υπέρ, 23 κατά. διαγράφεται αυτή η παραγραφός 5 από το συμβιβασμό, όπως προτείνεται. Και περνάμε λοιπόν στη συμβιβαστική D. Okay, we vote the compromise. Uh, συμβιβαστική με την διαγραφή τη. Όχι, όπως, το λέ, αναφέρεται στη συμβαστική πρόταση. Είναι σαφές Την παράγραφο 5. Παράγραφος 5. Υπέ. Όπως προτείνει λοιπόν η συμβαστική πρόταση σε σχέση με την παράγραφο 5. Ψηφίζουμε λοιπόν... We vote on the original as Ψηφίζουμε λοιπόν ε, όπως προτείνεται για την παράγραφο 5. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Νομίζω ότι θα πρέπει να ελέγξουμε το αποτέλεσμα έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Υπέρ. Κατά. Μάλιστα. Έχουμε δύο ψήφους κατά. Επιπλέον. υπέρ της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. we go to compromise. Συμβαστική D λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική E. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική F. Υπέρ. Excuse me. Uh, excuse me, we vote amendment. Ψηφίσαμε την 243. Ε, ναι, ναι, ναι. Ψηφίσαμε την 243 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική F. Ευχαριστώ, Ζαν Πολ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στη συμβιβαστική G. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία, την 255. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Excuse me, point of... Ένα διαδικαστικό θέμα να θίξουμε. Απορρίφθηκε η παράγραφος, η παράγραφος 5 στη συμβιβαστική C. Θα πρέπει ξεχωριστά λοιπόν να ψηφίσουμε τις τροπολογίες. Όλες ε, αφορούν την ε, διαγραφή, αλλά την 194 την 194 πρέπει να την ψηφίσουμε παρόλα αυτά. Στην ε, τέταρτη σελίδα. Η 194, επειδή διαγράφει παράγραφος 5, θα πρέπει αυτές οι τροπολογίες που αφορούν τον παράγραφο να ψηφιστούν ξεχωριστά. Η μία όμως δεν αφορά διαγραφή. Η 194 αφορά την διαγραφή. Ψηφίζουμε την 194. Είναι σαφές. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και πολύ λυπάμαι για την ε, σύγχυση και πάλι περνάμε στη συμβιβαστική age. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Συγγνώμη, έχετε δίκιο. Ψηφίζουμε τις αιτιολογικές ε, σκέψεις. 54, Τραπολογία 54, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55, υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 56, υπέρ, κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θα μπορούσαμε να ελέγξουμε την 55. Την 55 ή την 56. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 56. τη Α, εγκρίθηκε η 56, είναι σαφές. Άρα, ε, λυπάμαι να ψηφίσουμε. Μήπως θα μπορούσατε να διευκρινίσετε κατά πόσον οι 55 και 56 εγκρίνονται και οι δύο σας παρακαλώ. Η 56 εγκρίθηκε, η 55 ε, δεν εγκρίθηκε. Νομίζω ότι ήταν η ίδια, ε, οι ίδιοι ψήφοι, λέει ο κ. Σβέν Κιγκόλτ. Εσείς ήσασταν υπέρ, όχι, το ΕΛΚ. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε για την 55. Ναι, να ελέγξουμε την ε, τροπολογία περιθμών 55 τότε. Την 55 ηλεκτρονικά. 55. What we Electronic against and then you vote. Ψηφίσατε, ψηφίσατε παρακαλώ. Την 55 σας παρακαλώ. Ψηφίσατε, Σβέν, εσείς υπέρ, μάλιστα. Η υπερβάνους ψηφίζει κατά. Ωραία. Πέρα ψηφοφορίας απορρίπτεται. Πολύ ωραία. Απορρίπτεται 55, εγκρίνεται 56 και τώρα περνάμε στη συμβιβαστική age. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. <coughs> Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα, παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. Όχι. Η Βάνς είναι υπέρ και ο Σβένιν είναι υπέρ. Άρα 23 ψήφοι υπέρ, 22 κατά, άρα εγκρίνεται και περνάμε στη συμβαστική ΑΗ τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική G. J. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική K. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L. Σε τμήματα. Ζητάει το L. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Και περνάμε έτσι στη συμβαστική M. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Συμβιβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική O υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική P υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q σε τμήματα έχουν ζητήσει οι σοσιαλιστές σε τρία τμήματα συγκεκριμένα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, Άποχες. Εγκρίνεται. Θέλετε να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Μάλιστα, το πρώτο τμήμα της συμβαστικής Q. Ελέγχουμε. Ε, Αν ψηφίσατε όλοι, έχουμε δύο επιπλέον ψήφους κατά. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε και το δεύτερο τμήμα, παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Οι υπερβάντς και ο Σβέν ψηφίζουν υπέρ. One in favor, one against. We close the votes. Μία μία κατά. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Υπέρ, τρίτο τμήμα, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στη συμβαστική R. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική S. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική T. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική V. U. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική V. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική W. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική X υπέρ σε δύο τμήματα. Ε, compromise X is... Ε, Η συμβαστική X ε, έχει δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της συμβαστικής X υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής 6. Two more, uh, negative votes. Δύο επιπλέον ψήφοι κατά. Σας παρακαλώ ψηφίστε όλοι. A few more is close. Πέρασε. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία Y. Ο κύριος Γκοζές. Νομίζω ότι οι φίλοι μας οι σοσιαλιστές παρουσιάζουν μία ψήφο επιπλέον από την αρχή της ψηφοφορίας. Μπορούμε να δούμε ακριβώς ποια είναι η σύνθεση της Επιτροπής μας αυτή τη στιγμή. Η Γραμματεία θα μετρήσει τους παρόντες. Νομίζω ότι δεν ισχύει, αλλά ούτως ή άλλως ζήτησε από τη γραμματεία να το ελέγξει. Ζήτησε και από τη δική μας γραμματεία να ελέγξει ότι δεν έχουμε ένα παραπάνω.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 So there are, uh, one more socialist, but not voting because... Υπάρχει ένας επιπλέον σοσιαλιστής όντως, ο οποίος δεν ψηφίζει όμως. Ό,τι πείτε εσείς κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Γκοζές. Πάντως νομίζω ότι και η ίδια συσκευή καταμετρά σωστά τον αριθμό. η συσκευή και η γραμματεία μας λένε τα πράγματα είναι εντάξει. Επομένω αυτό δεχόμαστε ως ε, πόρισμα. Άρα συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Μάλιστα, συνεχίζουμε στην συμβαστική τροπολογία Y, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική Z σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική διπλό α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AE υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51. Κυρία Κλέβε, θέλετε το λόγο. Δώσουμε ψηφοφορία και θα πάρει το λόγο αμέσω μετά. Τροπολογία 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το κείμενο συνολό το τροποποιήθηκε υπέρ. Η κυρία Κλέβα θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ένα πράγμα μόνο θέλω να πω. Θα ήθελα επεξήγηση ψήφου εξ ονόματος των ε, σοσιαλιστών. Ε, Εξαιτία τη ε, πάρα πολύ καλή έκβαση τη ψηφορία για την τροπολογία τη συμβαστική ΣΥ, θα ήθελα να πω στην πολιτική μου ομάδα να ψηφίσει υπέρ τη έκθεση αυτή και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την γνωμοδότησή του αυτή και για όλε τι απόψει τι οποίε δέχτηκε του τελευταίου 4-5 μήνε που συζητάμε την έκθεση αυτή Εργαστήκαμε πολύ σκληρά και προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε το ποσοστό 40% καθώς επίση και όλο το σύστημα κυρώσεων το οποίο προβλέπεται. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Κλέβα. Ψηφίσουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικός. Πέρας. 37 υπέρ, 39 μάλλον υπέρ, 2 κατά, 6 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Όλε Σμιτ. Λύεται συνεδρίαση και θα τα ξαναπούμε σήμερα το απόγευμα στις 3.